Señor Presidente. Muy buenos días. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Άρχεται η Σύνοδος. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω θερμά στην αίθουσα